και θα δούμε κατά πόσο το εμπόριο με τις εκπομπές αυτές είναι ένας καλός δρόμος για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 12. Η επόμενη συνεδρία θα διεξαχθεί αύριο 5η